Θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι ο κύριος Φρανκ Βαν Χέκε προσχώρησε στην Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Δημοκρατίας με ισχύ από την 9η Νοεμβρίου 2011. Υπογραφή πράξεων που υιοθετήθηκαν βάσει της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας την ε, Τετάρτη θα υπογράψω 16 τέτοιες ε, πράξεις σύμφωνα με τον κανόνα 74 του εσωτερικού κανονισμού.